Λοιπόν, συνάδελφοι και υπόλοιποι παρόντες, ας ξεκινήσουμε. not very many this afternoon, but it's quality. Δεν είμαστε πολλοί. Ούκεν το πολλό το F, όπως πάντα. Και χαιρόμαστε που είναι εδώ και ο annual. Uh, που παρουσιάζει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού, και, του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Αρκομανία και όλοι έχετε την έκθεση μπροστά σας, στο έδρανό σας, έκθεση του 2013 και online υπάρχουν κάποια διαδραστικά εργαλεία που συνοδεύουν την έκθεση που παρουσιάζουν μεγαλύτερες λεπτομέρειες σε συγκεκριμένα θεμάτων όπως χρήση κανάβεως υψηλού κινδύνου, χρήση του κοκαίνης σε, σε περιπτώσεις κινδύνου, ψυχοτροπικές ουσίες και υπατήτης γάμα για κάποιες συγκεκριμένες χώρες χωρίς χρονοτριβή. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Γκούτζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Είναι πράγματι μεγάλη χαρά για μένα για μία ακόμη φορά να είμαι εδώ μαζί σα και να μοιραστώ μαζί σα την ανάλυση του παρατηρίου όσον αφορά την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη για το 2013 και είμαι πολύ χαρούμενος διότι από τώρα και στο εξή μπορούμε να σας δίνουμε μια ανάλυση ένα εξάμεινο νωρίτερα από ό,τι μας ζητήσατε. Και αυτή η εξέλιξη είναι πραγματικά κάτι αναγκαίο για να μπορούμε να προσαρμοστούμε με τον ρυθμό αύξησης του φαινομένου του, των ναρκωτικών. Κάτι που ήδη ανέφερε η ανάλυση μας Έχουμε ένα πακέτο δηλαδή, ολοκληρωμένο. Και ελπίζω να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στι προσδοκίε των διαφόρων ακροατηρίων και ιδίω εκείνων που διαμορφώνουν την πολιτική. Λοιπόν, υπάρχουν και τα στοιχεία online που ίσως θα μπορέσουν να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες, αυτές που χρειάζεστε. Στο πίκε του πακέτου είναι η έκθεση με τι εξελίξει που έχετε μπροστά σα για τα ναρκωτικά Βλέπετε σύνοψη. and on Europe's uh, responses uh, to these developments. Και τι απαντήσει Ευρώπη στα διάφορα προβλήματα. Να πω μερικά λόγια για την ηρωίνη και τα οπιοειδή. Αν δει κανεί το όλο τοπίο των ναρκωτικών της Ευρώπης, πολλά ναρκωτικά που καθορίζουν τις τελευταίες δεκαετίες το πρόβλημα, είναι σταθερή κατάσταση και μειούται το πρόβλημα. Η ηρωίνη το ναρκωτικό που μακρόν ήταν στο επίκεντρο του προβλήματος φαίνεται να χάνει η ηρωίνη. Και αυτή η εξέλιξη έλαβε χώρα έναντι, έναντι δραματικής αυξήσεως στη θεσιμότητα της θεραπείας των ναρκωτικών και διάφορων υπηρεσιών που παρέχονται και παροχή με δράση που, ε, και η δράση προσπαθεί να μπλοκάρει τους δρόμους εισόδου στην Ευρώπη όσον αφορά τη θνησιμότητα ε, τα οπιοειδή και η ηρωίνη ε, οφείλουν δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα στην Ευρώπη ίσως να αλλάζει βλέπουμε διάφορους δείκτες και βλέπουμε να μειώνεται το φαινόμενο μειώνεται η νέα ζήτηση για θεραπεία για ηρωίνη ε, λιγότερο είναι χρησιμοποιείται μέσω ενέσεως γυράσκουν οι χρήστες και μειώνεται και ο αριθμός ε, θανάτων από υπερβολική χρήση. Και τα φαινόμενα καταληψίας που οφείλονται στη χρήση της ηρωίνης μειώνονται και μειώθηκε η προσφορά ηρωίνης. Θεραπεύονται περισσότεροι άνθρωποι. 730.000 ε, θεραπείες. 730.000 ε, άνθρωποι θεραπεύονται μέσω υποκαταστάτων της ηρωίνης. Και συνολικά για όταν ναρκωτικά 2 εκατομμύρια ασθενείς θεραπεύονται. Η μεθαδόνη χρησιμοποιείται κυρίως σαν υποκατάστατο και η προπιονοφήνη χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο πάνω από 50% των χρηστών ηρωίνης στην Ευρώπη ε, τελούν υποθεραπεία με υποκατάστατα. Αυτό είναι υποφελές για την υγεία τους. Αλλά μειώνεται και το έγκλημα που σχετίζεται με τη χρήση ναρκωτικών. Και μειώνεται και η ζήτηση. Επενδύσεις για θεραπεία πρόληψη και μείωση βλαβών σημαίνει ότι έχει προχωρήσει η Ευρώπη και μειώνεται ο κίνδυνος όσον αφορά τη μόλυνση από AIDS λόγω χρήσης ναρκωτικών μακροπρόθεσμα. Βλέπουμε μείωση στην Ευρώπη των νέων μολύνσεων από το AIDS από το 2004. Από το 2011 είδαμε να διακόπτεται η προς τα κάτω πορεία. Μια μικρή αύξηση βλέπουμε. Νέες μολύνσεις. Κυρίως σε προβλήματα και ξεσπάσματα των προβλημάτων στην Ρουμανία και την Ελλάδα. Έχουμε και την κρυπτοεπιδημία υπατήτηδας γάμα από εκείνους που χρησιμοποιούν τα ναρκωτικά μέσω ενέσεων. Ε, ο κόσμος πολύ συχνά δεν ξέρει ότι έχει αυτό το πρόβλημα. Και αν δεν θεραπευτούν, η ασθένεια αυτή μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγείας και θάνατο. 18 με 80% από τους που χρησιμοποιούν ενέσεις ε, μολύνονται από τον ιό ανάλογα με τη χώρα. Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ διότι υπάρχουν θεραπείες για την υπατήτη γάμα που, που διατίθενται όλο και ευρύτερα για την κάναβη. Χρησιμοποιείται ευρύτατα. Και είναι και επίμαχο ναρκωτικό. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την ε, προμήθεια κανάβεως στην Ευρώπη. Ε, λόγω των αλλαγών στον τομέα των συνθετικών ναρκωτικών. Θέλουν οι παραγωγοί να είναι εκείνοι που παρέχουν τα ναρκωτικά να είναι πιο κοντά στους καταναλωτές. Έχουμε τη μαριχουάνα και χασίσει Αυτές οι δύο μορφές της κανάβεως. Ε, η μαριχουάνα είναι πιο διαθέσιμη, περισσότερο διαθέσιμη. Το 2010 είχαμε περισσότερες κατασχέσεις ε, μαριχουάνας από ότι ε, οποίου a on the balcony to major production sites. Λοιπόν, η παραγωγή της κανάβιος ε, είναι ιδιαίτερα προβληματική. Έχουμε συμμορίες εγκληματικές και υπάρχει και η δυνατότητα βίας, ξέσπασμα βίας και σε σχέση με άλλα ναρκωτικά και παράνομα ναρκωτικά και εγκλήματα. Η κανάβις χρησιμοποιείται περισσότερο. 77 εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το ναρκωτικό σε κάποια φάση της ζωής τους. 15,4 εκατομμύρια νέοι ενήλικες ε, είναι χρήστες και αναφέρθηκαν τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή ε, νοούμε 15 με 34 ετών. Πάνω από 3 εκατομμύρια καθημερινοί χρήστες, ε, νέοι άντες κυρίως, χρησιμοποιούν την κάναβη και βλέπουμε πιο πολύ είναι υπόκειται στη θεραπεία που προβλήμα δημιουργεί η κάναβης και πολλοί πηγαίνουν για πρώτη φορά για θεραπεία και είναι χρήστε κανάβιους. Οι περισσότερε αλλαγέ. είναι περίπλοκο και δυναμικό το πρόβλημα των ναρκωτικών και δημιουργεί πολλές ε, προκλήσεις. Για πολλαπλούς λόγους χρησιμοποιούνται ναρκωτικά. Δύσκολο να λύσει το πρόβλημα κανεί επικοινωνόμενο σε ένα ναρκωτικό, κυρίω στα χημικά. Οι χρήστε χρησιμοποιούν χάπια, σκόνη, ανάλογα με αυτό που βρίσκουν. Και ανάλογα με την ποιότητα που θεωρούν. Η κοκαίνη χρησιμοποιείται περισσότερο. 2,5 εκατομμύρια νέοι χρησιμοποίησαν το ναρκωτικό τελευταίο χρόνο. Για τα διάφορα ασθεντικά ναρκωτικά, έκσταση 1,8 εκατομμύρια, αμφεταμίνη 1,7 εκατομμύρια, Μιλάμε για τους νέους πέρσι, τη χρήση κάνουν. Το πιο δημοφιλές, <coughs> ναρκωτικό ποικίλει από χώρα σε χώρα. Στη Βόρεια Ευρώπη χρησιμοποιούνται περισσότερο εμφεταμίνες. Και στο Νότο, η κοκαίνη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το 2008 είχαμε την ανώτατη χρήση της κοκαίνης και μετά έχουμε μείωση Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιείται περισσότερο. Σε άλλε χώρε με μικρότερη χρήση δεν βλέπουμε παρόμοιε αλλαγέ, σημαντικέ αλλαγέ, σχετικά σταθερή χρήση. Βλέποντα την αγορά, από το 2008 μειώθηκαν οι κατασχέσει. Έχει μειωθεί και η ζήτηση. Οι ποσότητε κοκαίνη μειώθηκαν το 2006. Κατά τη διάρκεια της περίοδου που πέρασε ε, μειώθηκε κατά το ίμιση η κατάσταση κοκαίνης. Έχουμε συγχυτικές εξελίξεις στις μεθαμφεταμίνες που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Σε περιορισμένο βαθμό χρησιμοποιήθηκε στην Ευρώπη μόνο στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Οι μεθαφεταμίνες χρησιμοποιούνται περισσότερο, είναι διαθέσιμες στην αγορά όχι πολύ σε όγκο, σε σχέση με άλλα ναρκωτικά. Εδώ χρειάζεται επαγρύπνηση. Οι μεθαμφεταμίνες μπορούν να διαδίδονται πολύ γρήγορα και να έχει πολύ ανεδική επίδραση στην υγεία. Γενικές εξελίξεις. Η καινοτομία επηρεάζει την εξέλιξη και η αύξηση της παραγωγής των θετικών αγορών και δεν, δεν σε κάποιο βαθμό η επιχειρήση κατά και κατάσχεση προδρόμων ουσιών έχει παίξει ρόλο, είναι σημαντικό. Είναι ένα παιχνίδι γάτας με το ποντίκι. Οι πρόδρομε ουσίε καλύπτονται από την νομοθεσία και για να βρουν την πρώτη, για να βρουν την πρώτη ύλη δυσκολεύονται όλο και περισσότερο. Όπω στον τομέα τη έκσταση. Η κατάσχεση χαπιών με το MTMA ε, μειώνεται λόγω προσπαθειών της αστυνομία που κυνηγούσε την πρόδρομη ουσία PMK. Αυτό επηρέασε και τη χρήση. Έχουμε όμως μία ανάκαμψη σκόνες με πολύ MTMA, διότι οι παραγωγοί μπορούν να παράγουν συνθετικά τις πρόδρομες ουσίες που απαιτούν. θα δούμε εάν αυτό οδηγήσει σε αύξηση του ενδιαφέροντος ο πλευράς νέων ή τη χρήση του ναρκωτικού στο μέλλον. Η πιο σημαντική εξέλιξη που βλέπουμε, που αποτελεί πρόκληση. Οι νέες ψυχότροπες ουσίες. Καμιά φορά εμφανίζονται στην παράνομη αγορά αυτές οι ουσίες και καμιά φορά σαν νόμιμες εναλλακτικές για τον έλεγχο των ναρκωτικών πολλούνται και καταναλώνονται παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για το πώς ασφαλείς είναι οι ουσίες. Πέρσι, το σύστημα αγκαίας προειδοποίησης έλαβε, χώρα, έλαβε γνώση για 73 νέες ουσίες. Από και συνολικά 280 ουσίες ανοιχνεύονται το σύστημά μας. Όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των, των ουσιών που εντοπίζονται είναι από πιο σκοτεινές ομάδες ουσιών εμφανίστηκαν νέα συνθετη, νέες συνθετικές ουσίες, καλαμινοειδή, που ε, και καφενώνες που ε, τα πρώτα πολλούνται σε υποκατάστατα της κανάβεως. Τελευταίο εννιάμινο κάναμε ανάλυση κινδύνου. Για, το, για ναρκωτικά πολλούνται σαν αμφεταμίνη και το 5AT, περίπλοκο χημικό, το προηγούμενο ήταν 5MA. Το δεύτερο πωλείται ως νόμιμο προϊόν. Πάνω από 40 νέοι έχουν πεθάνει ε, λόγω χρήσεως αυτών των δύο ουσιών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Οι νέοι έχουν γίνει ε, ε ζωά, σαν ζωά, στα οποία, σαν πειραματόζα, στα οποία δοκιμάζουν η παραγωγή ε, νέες ουσίες. Μέχρι τώρα οι χώρες Κάνουν πειράματα με διάφορα μέτρα ελέγχου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Τρεις βασικές προσεγγίσεις ήταν η νομοθεσία, θέσπιση νέων νόμων με βάση τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες ή άλλα είδη ελέγχων, φάρμακα και νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτών. Χρειάζεται πρόληψη και μείωση κινδύνου με σχετικές στρατηγικέ. Να κινούμεθα ταχύτερα. Να μπορούμε να τοπίσουμε ταχύτερα και τα αποκρινόμεθα σε συγκεκριμένε επικίνδυνες ε, ουσίες και προϊόντα. Χρειαζόμαστε λοιπόν το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση ε, που πρέπει να λειτουργεί καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει πρόταση για νομοθετησία για να ενισχύσει το μηχανισμό. Κλείνοντας, να αναφέρω το πλαίσιο για την στρατηγική για τα ναρκωτικά. Το τοπίο έχει αλλάξει λόγω παγκοσμιοποίησης και τεχνολογικής καινοτομίας και λόγω, πειραμα... λόγω μειώσεως πειραματικής χρήσεως μένουν αυτοί που χρησιμοποιούν τα ναρκωτικά μόνιμα. Όλα τα αναφερθέντα. Και αυτοί αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, ε, ε, οι πιο μόνιμοι χρήστες. μπορούμε να είμαστε γέννη αισιόδοξοι. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την μείωση της ζήτησης δίνουν καρπούς. Θα μειώσουμε προσφορά και τη ζήτηση. Είχαμε αποτελέσματα, αλλά απομένουν πολλά προβλήματα παλιά και καινούρια. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Κυρίως τώρα που η καιρή είναι πολύ χαλεπή από οικονομικής πλευράς για πολλές χώρες. Η ανάλυση παρουσιάστη στην έκθεσή μας δείχνει ότι μπορούμε και πρέπει να ανταλλάξουμε εμπειρίε να μάθουμε ένας τον άλλον, μόνο με συντονισμό και συνεργασία θα είναι αποτελεσματικά τα μέτρα μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τον επόμενο μήνα θα λάβετε την Γενική Έκθεση Δραστηριοτήτων. Θα αφορά το 2012. θα υιοθετηθεί σύντομα και στις 15 Ιουνίου θα παραδοθεί το αργότερο. Και αν θέλετε να σας τη στείλω, ειδοποιήστε με παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκούτζ. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Και εγώ θέλω να μιλήσω. Κυρία Γομέρο Λόπες, μετά η κυρία Σίπουλ και μετά η κυρία Μόρβαη, η κυρία Ρομέρο πρώτη. Gracias, Presidenta. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την παρουσία του Διευθυντού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ναρκωτικών, η παρουσία του εδώ είναι σημαντική όπως και η έκθεση η οποία ήταν ε, είναι πιο προσαρμοσμένη στους καιρούς από τις προηγούμενες ε, παρουσιάσεις που μας δίναν στοιχεία τα οποία δεν ήταν τόσο ενημερωμένα. Η δική του παρουσίαση είναι επικαιροπεμένη και, έχει... και είναι σημαντική για μας. Εγώ συμμερίζομαι το, το ότι το θέμα των ναρκωτικών στην κοινωνία μας είναι θέμα δημόσιας υγείας. Αφορά την υγεία των συμπολιτών μας. Και ίσως ε, θα έπρεπε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε οτιδήποτε αφορά το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, όπως άλλωστε και για την εμπορία ανθρώπων. Αυτό το παρατηρητήριο μάλλον θα έπρεπε να αφορά περισσότερο την δημόσια υγεία των πολιτών και όχι τόσο τα φαινόμενα του εμπορίου, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο η προσοχή μας ε, στο θέμα αυτό, γιατί επιδεινώνεται η υγεία των πολιτών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε τις στρατηγικές των χωρών μελών, να δούμε ποιες χώρες είναι αυτές που πάσχουν περισσότερο από τις επιπτώσεις των ναρκωτικών και ποια θα ήταν τα πιο ενδεδειγμένα μέτρα καταπολέμησης αυτού του φαινομένου. Τα τελευταία χρόνια ε, τελικά έχουμε εξισώσει τους ε, μπόρους με τους ε, χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κατά την άποψή μου, όπως είπα, το παρατηρητήριο θα έπρεπε να επικεντρώσει την προσοχή του όχι τόσο στην εμπορία, αλλά στις επιπτώσεις των ναρκωτικών στην υγεία των πολιτών. Το πρόγραμμα της Κομισιόν και τα προγράμματα των χωρών έχουν αξιολογηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η επίπτωση αυτών των προγραμμάτων στον πληθυσμό. Ποια από αυτά τα προγράμματα είναι πιο αποτελεσματικά. Ποια είναι η επίπτωση σε πιο σκληρά ναρκωτικά όπως είναι η ηρωίνη για παράδειγμα ή σε πιο ήπιους τύπους ναρκωτικών. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να γίνει δηλαδή μια αξιολόγηση. Το δεύτερο αφορά τους θανάτους από υπερδόση, από υπερβολική δόση. Ε, η έκθεση λέει ότι υπάρχει μια μείωση των θανάτων. Γνωρίζετε γιατί υπάρχει αυτή η μείωση κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται εν μέρη στη μείωση της χρήση ηρωίνης. Αλλά επίσης ε, σχετίζεται και με αυτά τα προγράμματα μείωσης της ε, ζημίας στην ανθρώπινη υγεία. Τώρα, όσον αφορά τις νέες ουσίες, είναι προφανές ότι η παραγωγή των ναρκωτικών, οι κατασκευαστές ναρκωτικών ε, παράγουν ε, όλο ένα νέα ναρκωτικά τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατάλογο των γνωστών ουσιών. Αυτό το οποίο είναι παράλογο είναι ότι για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα ενός έτους. Ενώ αυτό θα μπορούσε να γίνει πολύ γρήγορα, μέσα σε μια μέρα ή δύο θα μπορούσε να εντοπιστεί και το νέο προϊόν και να συμπεριληφθεί άμεσα στον κατάλογο. Γιατί αλλιώς ε, στο διάστημα αυτό του ενός έτους θα υπάρξουν Πολύ θάνατοι από αυτές τις ουσίες. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζίπελτ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη που δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την παρουσίαση. Αλλά θα ήθελα να θέσω δύο ή τρία ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί και στο παρελθόν και τώρα αναφέρονται και στις, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι όλο και περισσότερο τα ναρκωτικά υποκαθίστανται από χημικά, συνθετικά ναρκωτικά. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσο αυτά τα χημικά, συνθετικά ναρκωτικά όσον αφορά την άμεση επίδρασή τους αλλά και το ζήτημα της μελλοντική εξάρτησης είναι ισχυρότερα από τα άλλα πιο φυσικά, φυσικής προέλευσης ναρκωτικά. Ε, αν υπάρχει μια τέτοια διαφορά ή όχι. Δεύτερον, ε, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι τα συνθετικά αυτά ναρκωτικά θα αντικαταστήσουν τα πιο συμβατικά ναρκωτικά ή θα αυξηθεί συνολικά ο όγκος των ναρκωτικών, θα προσθεθούν δηλαδή στα ήδη υπάρχοντα. Το άλλο ερώτημα είναι κατά πόσο θα πρέπει, ε, κατά πόσο αλλάζουν τα δίκτυα παραγωγής και διανομής αυτών των συνθετικών ναρκωτικών και κατά πόσο δεν χρειάζεται μια νέα μορφή συνεργασίας με τις αστυνομικές αρχές, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες ε, δομές ε, και οι νέοι δρόμοι των ναρκωτικών. Η κυρία Μορβάη, πολιτικός, πόσο η μεγαλύτερη πρόκληση και το πιο ενδιαφέρον ε, στοιχείο της έκθεσης είναι στη σελίδα 12 για την κάναβη είναι το ναρκωτικό που διχάζει την ε, ε, κοινή γνώμη. Κάποιες χώρες κάνουν σαφώς τη διάκριση ανάμεσα στην κάναβη αφενός και άλλες ναρκωτικές ουσίες ε, αφετέρου στην πολιτική τους για τα ναρκωτικά. Βάσει τη της έρευνας που έχει γίνει και των γνώσεων που έχουμε, τι πιστεύετε εσείς, είναι αυτό δικαιολογημένο, αυτή η στάση, αυτή η διάκριση. Ε, cannabis Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσέγγισεις για τη χρήση. Η φιλελεύθερη προσέγγιση, όπως αποκαλείται, βάσει της οποίας, ε, εντάξει, καλή είναι η κάναβη, δεν είναι επιζήμια για την υγεία, δεν προκαλεί εξάρτηση. Υπάρχουν ε, χώρες ε, που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, κανένα συμφέρον για να παρέμβουν σε σχέση με τη χρήση της. Στην Ουγγαρία, παραδείγματο χάρη, έχουμε ε, διασημότητες, δημοσιογράφους, μοντέλα, ακόμη και πολιτικούς, γνωστούς συγγραφείς που κάνουν χρήση δημοσίως χωρίς να το κρύβουν και μάλιστα αποτελεί και σημάδι απελευθέρωσης ε, ελευθερίας. Ε, και βλέπουμε στην έκθεσή σας ε, ότι υπάρχουν πολλαπλές προσεγγίσεις σε σχέση με τη χρήση της κάναβης στο κεφάλαιο που αναλύεται τις διαθέσιμες ιατρικές αγωγές. Και για τους εφήβους σας λάβουμε υπόψη ότι αυτό είναι κάτι καινούριο, δηλαδή αναρωτιούνται μα γιατί πράγμα μιλάνε, γιατί χρειαζόμαστε ιατρική αγωγή για την κάναβη. Ε, απλώς είναι ένα χαλαρωτικό, φυτικό, φυσικό προϊόν. τι, τι είδους προβλήματα υγείας μπορεί κάποιος να αναπτύξει με τη χρήση κάναβης και γιατί να χρειάζεται ε, ιατρική παρακολούθηση αγωγή ε, Πού βρίσκονται οι έρευνες, τι ξέρουμε για την κάναβη, τι ξέρουμε για τα, ε, τον αντίκτυπό της επί της ε, σωματικής και πνευματικής υγείας. Και τι πιστεύετε για αυτές τις δύο προσεγγίσεις για τα μαλακά και τα σκληρά ναρκωτικά. Είναι δικαιολογημένη όχι από ιδεολογική σκόπια, ε, ε επί τη βάση των γνώσεων που έχουμε στο στάδιο που βρίσκονται τώρα οι έρευνες. Ε, η κυρία Ιντβέλντ, ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω και εγώ τις τελευταίες ερωτήσεις, άμα δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Ε, εν μέρη με πρόλαβε η κυρία Μόρβαϊ. Μία από τις χώρες που ακριβώς έχουν διαφορετική πολιτική ε, σε σχέση με τη χρήση κάποιων ε, ειδών κάναβης ε, είναι η Ολλανδία. Φυσικά δεν είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε κυρία Μορβάη, είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Πρόσφατα ε, έγινε πιο αυστηρή, έγινε πιο αυστηρή η πολιτική μας για τα διάσημα coffee shops ε, είδαμε ότι ακόμη και τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα είναι μάλλον καταστροφικά. Αυξάνεται η χρήση, μειώνεται ο έλεγχος, ε, έχει ξανακυκλοφορήσει στους δρόμους και στα χέρια των εγκληματιών αυτό το ναρκωτικό και τελικά ε, αποφάσισαν όλοι ότι η αναθεώρηση πολιτικής δεν βοήθησε και πολύ. Αλλά σίγουρα δεν προωθείται η χρήση με την πολιτική μας. Να σας ε, μιλήσω επίσης ε, για ε, αυτό το φοβερό νέο ναρκωτικό που χρησιμοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και που σχετίζεται, από ό,τι φαίνεται, με την κρίση και την φτώχεια που πλήττει την Ελλάδα. Φαντάζομαι δεν το έχετε ακόμη συμπεριλάβει στην έκθεσή σας, γιατί φαίνεται να είναι πρόσφατη η εξέλιξη. Και η δεύτερη ερώτηση, ε, στον απόϊχο της φαρέμας, κυρία Δρομέρο, εσείς συντάσσετε την ετήσια έκθεση και εμείς θέτουμε την ετήσια ερώτηση. Καταμετρήσατε τον αντίκτυπο των διαφόρων πολιτικών για να δείτε πώς επηρεάζονται οι χώρες, οι διάφορες χώρες, οι διάφορες πληθυσμιακές ομάδες και σε σχέση με διάφορες κατηγορίες ναρκωτικών. Εντάξει, η χρήση ναρκωτικών είναι κάτι ε, ε, απευκταίο, αλλά πρέπει να ξέρουμε και ποιο είναι ο αντίκτυπος των πολιτικών. Ένα... Θα σας ζητήσω λοιπόν να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, αλλά θα φανώ λογικός. Κυρία Ρομέρο Λόπες. είναι κυρίως πρόβλημα υγείας, μας είπατε, το πρόβλημα της ε, κατάχρησης ναρκωτικών. Αυτό το βλέπουμε στην πλειοψηφία των κρατών μελών. Αν δείτε πώς γίνεται ο συντονισμός διαφέρει από χώρα σε χώρα και τα τελευταία δέκα χρόνια έχει περάσει το πράγμα από τη σφαίρα της επιβολής του νόμου στη σφαίρα της δημόσιας υγείας ε, αλλά ε, στην πλειοψηφία των κράτων μελών. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σας πω ότι πάντοτε θα πρέπει να βλέπετε τις δύο όψεις ε, του νομίσματος. Η εντολή μας είναι να καλύψει και την πτυχή επιβολής του νόμου σε σχέση με τα ναρκωτικά αναπτύσσουμε δείκτες ε, της ε, προσφοράς, παραδείγματος χάρη. Τυποποιείται η υποβολή εκθέσεων για να παρακολουθούμε την προσφορά. Ε, αν μπείτε σε περισσότερε λεπτομέρειες στου αρμόδιους οργανισμούς θα δείτε ότι τουλάχιστον 80% του προσωπικού ασχολείται με το θέμα υγείας και το 20% ασχολείται με το θέμα της μελέτη τη προσφορά και των τάσεών τη. Με ρωτήσατε αν γίνονται αξιολογήσεις ε, των πολιτικών. Ε, ναι, και τώρα θα συνδέσω το δικό σα ερώτημα με αυτό της κυρίας Ίντβελ. Δεν έχουμε ε, εντολή για να αξιολογούμε τι εθνικέ πολιτικές. Το Κοινοβούλιο, όταν έγινε η αναθεώρηση του κανονισμού την 1η η του 2007, το Κοινοβούλιο επιθυμούσε να μας δώσει εντολή και για την αξιολόγηση των πολιτικών, αλλά είναι προφανές ότι δεν το επιθυμούσαν τα κράτη-μέλη και αυτή τη στιγμή ε, η εντολή μας σταματάει σε αυτό το σημείο δηλαδή ανάπτυξη εργαλείων αυτοαξιολόγησης για τα κράτη-μέλη. Εμείς πάντως δεν ε, κάνουμε αξιολόγηση των πολιτικών, αξιολόγηση των μέτρων που αναλαμβάνονται κάνουμε και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι τη δουλειά μα. Η διάδοση των πληροφοριών είναι σημαντικό. Έχουμε το, πόρταλ, τη δικτυακή πύλη για τις βέλτιστες πρακτικές στον ιστότοπό μας και βλέπετε ε, εκεί πληροφορίες σε σχέση με τι λειτουργήσε και τι δεν λειτουργήσε σε ορισμένες συνθήκες από πλευράς πολιτικής και μέτρων τα κράτη-μέλη αλλάζουν ορισμένες φορές ε, την ε, πολιτική τους, μας ζητάνε ακόμη και σε εμπιστευτική βάση εξειδικευμένε ε, συμβουλές είτε μιλάμε για κοινωνική ένταξη, για τα καταπολέμηση της χρήσης, πάντοτε κάθε μέτρο το εξετάζουμε σε συνάρτηση με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και σε συνδυασμό με τη Γενική Έκθεση ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να αποκομίσουν τα στοιχεία που του τα ενδιαφέρουν. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή όμως να σας πω ε, ε, να σας δώσω νούμερα για την παραγωγή κάναβης ή άλλων ναρκωτικών αναχώρα. Δεν έχω τα πετούμενα στοιχεία μαζί μου. Για την πρόληψη ήταν το επόμενο σημείο. Σημειώθηκε βελτίωση βελτίωση ε, ε, χάρη κυρίως της ε, θεραπείας αντικατάστασης της ερωίνης. Η ναλοξόνη που είναι ε, κάτι που βοηθάει σε περίπτωση overdose, υπερβολικής δόσης ναρκωτικών. Εάν κάποιος διακομιστεί εγκαίρως στο νοσοκομείο και λάβει αυτή την ουσία, ε, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα καταφέρει. Οι χρήστες ηρωίνη ε, που βρίσκονται σε οικογενειακό περιβάλλον ή σε κάποιο συγκεκριμένο περιβάλλον μπορούν να κάνουν τη χρήση αυτής της ουσίας. Φίλοι ε, ή συγκάτοικοι μπορούν να προμηθεύουν στο χρήστη ε, ποσότητες αυτού του, αυτής της ουσίας αντικατάστασης. Γίνονται πολλέ δοκιμές και σε ορισμένε περιπτώσει θα αναφερθώ μόνο σε μία, ε, εξαιρετικά ε, επικίνδυνη περίοδος είναι ε, μετά τον, τη φυλάκιση όταν κάποιος βγαίνει από ένα σοφρονιστικό ίδρυμα και έχει ευκολότερη πρόσβαση σε ναρκωτικές ουσίες κυρίως άνθρωποι που για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουν κάνει χρήση ηρωίνης εύκολα ε, πέφτουν σε αυτή την παγίδα στις φυλακές. Δεν υπάρχει αρκετά ε, ε, στενή παρακολούθηση τόσο ώστε να χρησιμοποιηθεί η ουσία αντικατάστασης. Η μείωση των, υπερβολικών, των περιπτώσεων υπερβολικών δόσεων δεν σχετίζεται με την προσφορά αλλά με την ελαχιστοποίηση των επιζήμιων συνεπειών. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για ένα μόριο συνθετικό που πρόκειται για, συνήθως για παράνομες, ε, ε, νόμιμες ουσίες. Ε, δεν, αυτή η ουσία δεν είναι σε, ένα κατάλογο εθνικό ή, κατάλογο του ΟΗΕ. Είναι μια νόμιμη ουσία και πρέπει να έχετε αποχρόντα λόγο για να εξετάσετε αυτή την ουσία και αυτό, αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε και είναι μεγάλο μείον για τον οργανισμό μας και ίσως όταν συζητηθεί μελλοντικά η αναθεώρηση της πολιτικής για την αξία αξιολόγηση για την έγκαιρη προειδοποίηση για τις ε, ε, ψυχοτρόπες ε, ουσίες θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κεντρικός χώρος αποθήκευσης όλων των ουσιών που βρίσκονται στην αγορά που δεν μπορούμε να πούμε ότι με το που προκύπτει ένα νέο μόριο θα ε, απαγορευθεί αυτόματα γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για παραγωγή ε, φαρμακευτικών σκευασμάτων ή για ε, προϊόντα καθαρισμού, οτιδήποτε. Άρα χρειάζεται συνεργασία και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Μόλις μαθαίνουμε ότι συνδέεται με ένα συγκεκριμένο κίνδυνο μία ουσία, με τη Europol κάνουμε μία κοινή έκθεση και συνήθως μας ζητάνε αξιολόγηση κινδύνου μπορεί αυτό να κρατήσει αρκετούς ε, μήνες, ε, ε, όπως συμβαίνει ούτως ή άλλως ανά τον κόσμο, αλλά δεν, μπορούμε. Πρέπει όμως να προχωρούμε πάρα πολύ γρήγορα. Ε, Βεβαίω πρέπει να λάβετε υπόψη ότι γίνονται περίπου 25 δοκιμέ αναουσία και δεν νομίζω ότι μπορεί ένας οργανισμός να κινηθεί ταχύτερα. Can I continue in English? Uh, for Mrs. Sippel, the uh, <clears throat> uh, general... Ε, τα ε, συνθετικά ναρκωτικά μας ε, ρωτήσατε ποιος είναι ο αντίκτυπος τους. Είδατε ότι έχουμε 5-6 διαφορετικές κατηγορίες συνθετικών ουσιών, αλλά στο εσωτερικό κάθε κατηγορία μία μικρή αλλαγή σε ένα μόριο μπορεί να έχει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Το 4-MA είναι ένα είδος αμφεταμίνης είμαστε πεπισμένοι ότι κατά λάθος ε, παρήχθη αυτή η ουσία γιατί όπως ε, και η αμφεταμίνη ε, δεν, μάλλον τίθεται σε εμπορία ω αμφεταμίνη και όχι ω μια διαφορετική ουσία και μάλλον αυτοί που το παρήγαγαν δεν ήξεραν και οι ίδιοι ότι πρόκειται για μια νέα ουσία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την κάναβη, παραδείγματο χάρη, έχουμε από τις 75 νέες ουσίες πέρσι 35 σχετίζονται με την κάναβη αλλά δεν μπορούμε να, ε, κάνουμε, να ταξινομήσουμε τα αποτελέσματα ανά ε, νέο προϊόν. Ε, Ποιε είναι οι γνωστές ε, και οι παλιές ουσίες, οι άλλες νέες που προστίθενται στις παλιές. Μπορούμε να σας πούμε ότι, όπως σας είπα και νωρίτερα, πως στις παλιές ουσίες, ε, ηρωίνη, κοκαίνη και κάναβη, είναι μάλλον σταθερή η πορεία ή και φθήνουσα. Αυτά είναι τα καλά νέα. Ε, τώρα, από πλευράς νέων ε, ναρκωτικών ουσιών, δεν μπορούμε να βασιστούμε ε, σε στατιστικά στοιχεία που δεν υπάρχουν. Θα λέγαμε ότι ε, μειώνεται μάλλον η χρήση, δεν διωγγώνεται το πρόβλημα στην Ευρώπη. Ε, τρόπον να το έχουμε υποέλεγχο, αλλά από την άλλη πλευρά γίνεται πιο δυναμικό το φαινόμενο και εγκυμονεί νέους κινδύνους απρόβλεπτους γιατί δεν είναι νέοι. Η οδή πορείας τώρα, η διάδρομη εμπορία των ναρκωτικών. Αυτό γίνεται όλο ένα και περισσότερο παγκόσμιο ζήτημα. Με τη Europol συνεργαζόμαστε στενά, με τη CIPOL για την κατάρτιση των αστυνομικών, ε, με τον ΟΗΕ, με την Παγκόσμια Ένωση Τελωνίων, με τη ΣΥΠΑ, με τους δρόσους, με την Αυστραλία. Ε, συνεργαζόμαστε όλοι, αλλά πάρτε το παράδειγμα αυτών των συνθετικών ε, ουσιών κάναβης ε, ε, που παράγονται στην Ινδία, στην Κίνα και στη συνέχεια έρχονται στην Ευρώπη. Δεν είναι αρκετά μεγάλος οργανισμός για να παρακολουθήσει όλους αυτούς τους διαδρόμους λαθρεμπορίου. και ε, πρέπει να ξέρετε ότι το λαθρεμπόριο γίνεται από κοινού με άλλα προϊόντα, άλλε ουσίες. Δεν είναι ποτέ μόνο τα ναρκωτικά. Ε, η κυρία Μορβάη, η διαφορά με ρωτήσατε ανάμεσα ε, στα μαλακά και στα σκληρά ναρκωτικά. Δεν χρησιμοποιούμε εμεί αυτούς τους όρους, διότι είμαστε πεπισμένοι ότι η ουσία είναι ένα στοιχείο, το αν είναι ή μάλλον ε, το ένα θέμα είναι αν είναι επικίνδυνη ή όχι ουσία, αλλά το άλλο ζήτημα είναι το μοντέλο χρήσης, κατάχρησης των ουσιών. Μπορείτε να πείτε ότι σε κάποιες χώρες ε, θεωρείται η κάναβη ε, μαλακό ναρκωτικό, αλλά με καθημερινή χρήση της κάναβης βλέπουμε διάφορες, διάφορα ψυχο ψυχοκοινωνικά προβλήματα λόγω της ε, ε, τακτικής καθημερινής ε, χρήσης της κάναβης. Δεν πρόκειται για αντικατάσταση όπως στην περίπτωση της ηρωίνης και αυτά τα 3 εκατομμύρια καθημερινών χρηστών είναι ανησυχητικό φαινόμενο. 77 εκατομμύρια έχουν χρησιμοποιήσει, έχουν κάνει χρήση μία φορά στη ζωή τους κάναβη ή κάποιο άλλο ναρκωτικό αλλά η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων που έκαναν χρήση μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές όταν περάσουν τα 30 το ξεχνάνε και είναι ένα επεισόδιο στη ζωή τους απλώς ε, ε, το πρόβλημα είναι η τακτική, καθημερινή χρήση ουσιών που ε, προκαλούν εξάρτηση. Η προσεγγίσεις δεν είναι και τόσο διαφορετικές από ε, χώρα σε χώρα στην Ευρώπη. Κάποιες έχουν πιο φιλελεύθερη πολιτική. Ε, για το ε, λαθρεμπόριο καμία χώρα δεν ακολουθεί φιλελεύθερη πολιτική. Έχετε επίσης κάποιες διαφορές ε, και είναι παράνομη η ουσία η κάναβη σε όλες τις χώρες. Εξάλλου υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές ε, σε σχέση με την αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων ανάλογα με την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας. Δεν είναι και τόσο μεγάλες οι διαφορές. Η χώρα που συνειδητά καθοδηγεί τους ανθρώπους προς το σύστημα υγείας είναι η Πορτογαλία. Όταν συλλαμβάνονται κάποιοι με μικρές ποσότητες παραδόσεις παραδείγματος χάρη αυτό το άτομο πρώτα ε, παρακολουθεί στα πλαίσια του συστήματος υγεία σε μία ενημέρωση και στη συνέχεια τον καθοδηγούν προς μία αγωγή ενώ στις άλλες χώρες ε, αυτό το ίδιο άτομο θα πήγαινε, θα εντασσόταν στο πλαίσιο της, της επιβολής του νόμου και όχι της ε, δημόσιας υγείας ε, αλλά από τη ΣΥΠΑ έρχονται οι πιο νέες εξελίξεις στην ιστοσελίδα ε, μας βλέπετε 11 διαφορετικές, 11 ε, ε, διαφορετικά θέματα που τονίζουμε. Σε σχέση με τις νέες προσεγγίσεις για τα ναρκωτικά κάνουμε επίσης σύγκριση ανάμεσα ε, στην ε, νομοθεσία που ισχύει στις ε, πολιτείες της Αμερικής σε σύγκριση με την Ουρουάη παραδείγματος χάρη η οποία αναθεωρεί την πολιτική της και σκέφτεται και το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης όχι της νομιμοποίησης, της νομοθετικής ρύθμισης της κάναβης γιατί το ίδιο ισχύει και για τον καπνό Πάντω Πάντως, ε, εμείς δεν γνωμοδοτούμε από αυτό γιατί είμαστε ε, κέντρο παρατηρητήριο ουσιαστικά. Ε, κυρία Ιντβέλτ, έφτασα σε εσά. ΣΥΣΑ ονομάζεται αυτή η ουσία στην Ελλάδα. Είναι μεθαμφεταμίνη. Το είπα και νωρίτερα, δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα γιατί είναι δύσκολο να ε, ε, καταλήξουμε σε στοιχεία. Είναι αμφεταμίνη και μεθαμφεταμίνη, ένα συνδυασμός των δύο στην Τσεχία και στη Σλοβακία υπάρχει μία ουσία που ε, πριν από ακριβώς 75 ε, χρόνια ε, έφτασε στην αγορά. Είναι υπερδιτίνη, ένα φάρμακο που χορηγείται ώστε να ε, γίνουν πιο δραστήριοι οι άνθρωποι, ε, κυρίως οι Ναζί στη Γερμανία το έδιναν στους ε, στρατιώτες και το γενικότερα χορηγείται στους στρατιώτες για να έχουν περισσότερο κουράγιο και χρησιμοποιήθηκε από το 1977, 1977 μέχρι το 1998 στην Ανατολική Γερμανία. Αυτή η υπερδιτίνη λοιπόν ε, στην ε, Τσεχία και στη Σλοβακία, αλλά κυρίως στην ε, Τσεχία ή στην πρώην Τσεχοσλοβακία τέλος πάντων, Ακόμη και σήμερα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η στην πρωην τσεχοσλοβακια τελος παντων ακομη και σημερα ειναι το μεγαλυτερο προβλημα η υπερδιτινη με μεθαμφεταμίνη είναι μία ουσία που δεν προκαλεί μόνο εξάρτηση όπως η αμφεταμίνη, αλλά καταστρέφει την προσωπικότητα ε, από ψυχολογικής και σωματικής πλευράς ε, στις ε, ΙΠΑ. Έχουμε δει συγκεκριμένες περιπτώσεις γιατί είναι εύκολη η παραγωγή αυτού του φαρμάκου. Αυτή η μεθαμφεταμίνη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ασία, στις ΙΠΑ, αλλά κυρίως στην Αυστραλία. Τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα, είναι κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει μόνο η υπερδιτή είναι ή μεθαμφεταμίνη σε σκόνη. Είναι σε πιο συμπυκνωμένη μορφή και ονομάζεται crystal meth. Ε, επίσης αποκαλείται. Είναι σε πιο συμπυκνωμένη, είναι σε κρυσταλλική μορφή και... Ε, ε, μπορεί κανείς να το καπνίσει. Αυτό δεν ισχύει για τη μεθαμφεταμίνη σε σκόνη. Ε, πάει κατευθείαν στον εγκέφαλο, δεν περνάει από ε, το στομάχι. Ε, και στη Γερμανία στη Βαυαρία και στη Σαξονία κυρίως όπου ε, λόγω της γεωγραφικής γειτνίας γιατί παράγεται στην Τσεχία αλλά και στη Σουηδία ε, ε, και στην Τουρκία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ουγγαρία έχουμε στοιχείο ότι κυκλοφορεί σε μεγάλες ποσότητες αυτή η ουσία και παράγεται όχι μόνο στην Τσεχία αλλά και στην Σουηδία, στη Λετωνία, Λιθουανία και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηλά στον κατάλογο είναι το Ιράν και η Νότια Αφρική από την πλευρά των των χωρών παραγωγών. Δεν είναι μεγάλες ποσότητες προς το παρόν, αλλά είναι ραγδαία η αύξηση των ε, ε, ποσοτήτων και είναι σοβαρότατα τα προβλήματα υγείας ε, με τη, μετά τη χρήση της ουσίας. Θα σταματήσω εδώ και αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν άλλα καυτά θέματα. Σύντομη παρακαλώ, συντομότατη. έχουμε πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η πρόταση της παρέμβασής σας ε, με κάνει να σκεφτώ αν να σας ρωτήσω αν ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο το οποίο να μπορεί να αξιολογήσει τις επιπτώσεις και να καταρτήσει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ίσως το παρατηρητήριο θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα τέτοιο κέντρο το οποίο να αξιολογεί τις επιπτώσεις αυτών των ουσιών και να μπορεί να θεσπίζει και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Ξέρετε, είμαστε ένας μικρός οργανισμός στην Ευρώπη, όπως σας είπα αλλά δεν έχουμε εργαστήριο, αλλά βεβαίως συνεργαζόμαστε με κάποια εργαστήρια και έχουμε και επίσης ε, στενή συνεργασία με ιατροδικαστικά κέντρα. Όπως σας είπα, η νομοθεσία αλλάζει και σύντομα η Επιτροπή θα παρουσιάσει ε, μια νέα νομοθετική πρόταση για αυτό το νέο μηχανισμό αξιολόγηση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να τον αναμένουμε, αναμένουμε αυτή την πρόταση της Επιτροπής. Νομίζω ότι θέλει να αποδώσει αυξημένο ρόλο στο κοινό ερευνητικό κέντρο. Αλλά αν με ρωτάτε άμεσα εμένα, εγώ λέω ότι αν είχαμε επιπλέον πόρους ε, θα είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε, αλλά δεν ξέρω. Ε, βρισκόμαστε σε εποχή περικοπών όπου κανείς δεν δίνει δεκάρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να, γίνει, να υπάρξει μια εξέλιξη. Ε, η Κομισιόν ε, καλείται να κάνει το σχεδιασμό. Ίσως το κοινό ερευνητικό κέντρο μπορεί εδώ να παρέμβει. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερής διάταξης. Okay, last um, Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σέγγεν. Χτες έγινε τριμερής διάλογος υψηλού επίπεδου για το πακέτο δικυβέρνηση Σέγγεν. Επετέφθη συμφωνία. Το πρωί η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων επιβεβαίωσε ότι συμφώνησαν κατά κράτη μέλη με το πακέτο όπω ε, ήταν το αντικείμενο διαπραγματεύση. Η κυρία Ράντα Βέμπερ, που ήταν η πραγματεύτριά μα, δεν μπορεί να παραστεί σήμερα, δυστυχώ. Και μου ζήτησε να διαβάσω μια σύντομη δήλωση που είναι η εξή. Είμαι ικανοποιημένη διότι μετά από σκληρέ και μακρέ διαπραγματεύσει και με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με τα κράτη-μέλη καταφέραμε, καταφέραμε αν θέλετε κουβεντούλε έξω παρακαλώ. Λοιπόν, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε σαφεί κανόνε μαζί με ελέγχου ε, και αποτίμηση των καταστάσεων και να εφαρμόζονται μέτρα έσχατη ανάγκη και να χρησιμοποιούμε ελέγχου σαν έσχατη ανάγκη στα εσωτερικά σύνορα Σέγγερ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνονται όποτε τέτοιε κρίσιμε καταστάσει προκύπτουν και αυτό ήταν στο επίκεντρο τη προσέγγιση που ακολούθησα όταν ασχολήθηκα με το ευαίσθητο αυτό θέμα. Πιστεύω στεναρά ότι η ελευθερία τη διακίνηση εντό των σύνορων του Σέγγεν θα πρέπει να διατηρηθεί και να είναι από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, ε, Επόμενο, θα καλέσω τον κύριο Κοέλιο, που είναι συγγητής για τον μηχανισμό αξιολόγηση Σέγγεν, να πάρει το λόγο και μετά όποιο άλλο θέλει να μιλήσει θα πάρει το λόγο. Και μπορεί και η Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, διαδικαστικά. Η έκθεση της κυρίας Βέμπερ για την τροποποίηση ε, του συστήματος αυτού Σέγγεν θα πάει στην Ολομέλεια. Η συμφωνία με το Συμβούλιο θα υποβληθεί ως τροπολογία στο, στην Ολομέλεια για να ολοκληρωθεί η συμφωνία πρώτης ανάγνωσης. Η έκθεση του κυρίου Κοέλιο απαιτεί κάποια άλλα βήματα στη ΛΥΜΠΕ διότι πρέπει να αλλάξει η νομική βάση. Και το κείμενο του συστήματος ο ΣΕΝΚΕΝ θα τροποποιηθεί δυνάμει το άθρο 70 της ε, συνθήκης που κανονικά δεν προβλέπει την εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Συμφωνήθηκε να διαβουλευτεί μαζί μας το Συμβούλιο, οπότε θα ξεκινήσουμε διαδικασία διαβουλεύσεων. Θα υποβληθεί το αίτημα από το Συμβούλιο για γνωμοδότησή μας. Ο uh, uh, κύριος Κοέλιο θα αναφέρει λεπτομέρειες και θα επανέλθω στην προθεσμία της τροπολογίας. Ας ακούσουμε τον κύριο Κοέλιο και οποιοδήποτε μέλη θέλουν να παρέμβουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε κάναμε μια συμφωνία με την Ελλανδική Προεδρία με μέρου του Συμβουλίου και ειλικρινά δεν είναι ακριβώς ε, η συμφωνία που θα θέλαμε εμείς από το Κοινοβούλιο, αλλά ανταποκρίνεται σε κάποιες ανησυχίες μας. Καταρχήν ενισχύει τη διακυβέρνηση του Σέγγεν και βάζει ένα τέλος στο καθαρά διακυβερνητικό σύστημα και δημιουργεί έναν ε, μηχανισμό ε, ε, δημιουργεί έναν ενισχυσμένο μηχανισμό που ασύστησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ρητά τη δυνατότητα να αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν διενεργηθεί παράνομοι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα μέσω μέσω της δυνατότητας επισκέψεων που δεν έχουν ε, προαναγγελθεί. Κατά την άποψή μου, τα βασικά επιτεύγματα είναι τα εξή. Καταρχήν, η ενίσχυση του οργανισμού της ε, η ενίσχυση του ρόλου συγγνώμη, της Επιτροπής που δεν ε, περιορίζεται μόνο σε ρόλο παρατηρητού. Το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα προηγείται διαβούλευση με το Κοινοβούλιο για κάθε πρόταση της Κομινισιών όσον αφορά το μηχανισμό εξέλιξης και το Κοινοβούλιο θα μπορεί να καλεί την Επιτροπή η οποία έχει ένα συντονιστικό ρόλο να απαντάει τις ερωτήσεις που ενδεχομένω υποβάλλει το Κοινοβούλιο και τέλος θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας και θα έχει πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά έγγραφα, όπως είναι τα κείμενα αξιολόγησης, τα κείμενα ανάλυσης των κινδύνων, τις ε, απαντήσεις των χωρών ε, μελών, τις εκθέσεις, παρακολούθησης και συστάσεις. Και αυτή, αυτό πραγματικά είναι ένα μείζον επίτευγμα, γιατί όπως γνωρίζετε στο παρελθόν, ε, δεν είχαμε καν αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης. Αυτές οι εκθέσεις αξιολόγησης θα βασίζονται σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση ε, και προβλέπουν την ε, συμμετοχή των θεσμικών οργάνων, αυξάνουν το βαθμό διαφάνειας, γιατί υπάρχει υποχρέωση να ενημερώνεται το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε σχέση με την αξιολόγηση των επισκέψεων και τη διατύπωση των συστάσεων και διατυπώνονται συγκεκριμένα μέτρα με χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή τους και προβλέπει ρητά η δυνατότητα αξιολόγησης εάν ε, έχουν γίνει παράνομοι έλεγχοι στα σύνορα και προβλέπει τη δυνατότητα να γίνονται ε, μη προαναγγελθήσεις ε, επισκέψεις και σε περίπτωση κάτι την υποχρεωτικό θα κοινοποιείται 24 ώρες πριν και θα ε, περιλαμβάνεται επίσης συνεργασία με την Frontex. Οι αξιολογήσεις θα γίνονται από μικρές ομάδες εμπειρογνωμόνων με την συμμετοχή της ε, Επιτροπής και έτσι ε, μπαίνει ένα τέλος στην ύπαρξη διπλών ε, διπλών ε, τρόπων αξιολόγηση. Θα υπάρξει ένας ενιαίος ε, μηχανισμός όλης της επικράτειας του Σέγγεν, όπου η αξιολόγηση θα γίνεται με έναν ενιαίο, ομοιόμορφο τρόπο. Και τέλος, θα δίνεται... θα δίνεται δυνατότητα συμμόρφωσης με τους κανόνες του Σέγγεν και δεν θα υπάρχει κανένα αίσθημα, θα πατάσετε κάθε αίσθημα ατιμορρησίας. Ε, θεωρώ ότι αυτός είναι ο θεμέλιος βράχος επί το οποίο οικοδομείται όλο το σύστημα του Σέγγεν. Η διασυνοριακή έλεγχη και ο ρόλος που έχουν εδώ οι χώρες μέλη θα διατηρηθεί και υπάρχει και το άρθρο 26 εναπόκειται σε, στην ε, ευχέρεια των κρατών να θεσπίσουν ή όχι ελέγχους, αλλά ε, μπορούν να... Αλλά πιστεύω ότι η οχι ελεγχους αλλα μπορουν αλλα πιστευω οτι η οποία έχει γίνει σε σχέση με τους φυστάμενους κανόνες του Σέγγεν είναι αρκετά μεγάλη, γιατί η έκφραση εκ μέρους των ε, πολιτών και το Κοινοβούλιο ε, και γίνεται σεβαστό το Κοινοβούλιο ως προς την ε, συμφωνία η οποία επετεύχθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας σε αυτό το θέμα και την εξαίρετη συνεργασία. Ένα τελευταίο σημείο. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας για τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη διαδικασία. Το Συμβούλιο υποσχέθηκε να διαβουλεύεται το Κοινοβούλιο έστω και αν αυτό δεν προβλέπεται από τη συνθήκη. Αυτό το οποίο είπατε πριν μου δώσετε το λόγο αλλά είναι προφανές ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα κάποιων διαπραγματεύσεων που έχουν προηγηθεί, ούτω ώστε για να, πετύχει, να φτάσει το πακέτο αυτό στην Ολομέλεια θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία διαβούλευση. Ω εισηγητή, συστήνω προ την Επιτροπή να δώσει ευνοϊκή γνώμη χωρίς, ε, στο κείμενο αυτό χωρί να προτείνει κάποιε τροπολογίε. Θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας, να έχουμε μια ταχεία διαδικασία και θα προσπαθήσω τις επόμενες μέρες να έχω ένα νέο σχέδιο σύνταξης και θα σας συστήσω την έγκριση του κειμένου και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε στη ΛΥΜΠΕ ή δυνατόν την επόμενη εβδομάδα ώστε το πακέτο αυτό να φτάσει στην Ολομέλεια ταχύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much and also... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας, τις δικές σας και της κυρίας Βέμπερ τα τελευταία χρόνια Ευχαριστώ για την υπομονή σας, την επιμονή σας, για το αποτέλεσμα που πετύχατε. Δηλαδή προτείνεται μια ιονή διαδικασία, πρώτη ιονή ανάγνωσης. Άντριου, κυρία Ντανούκα, ο κύριος Έντσου πρώτος. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συμμετείχαν στις συζητήσεις. Συνεργαστήκαμε με αυτούς. Υπήρξε μεγάλος, καλή συνεργασία. Ευχαριστώ τον Κάρλος και την Ρενάτε διότι ε, ήταν πολύ επιδέξει στους χειρισμούς τους στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Τέσσερα χρόνια κράτησαν οι διαπραγματεύσεις. Τόσο νομίζω ότι κράτησε η διαδικασία. Έχω το εξή να πω. Όπως γνωρίζουμε, δεν είναι η τέλεια συμφωνία κατά την άποψή μας, αλλά είναι μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση συγκρίση με την πρώτερη κατάσταση. Ο χώρος Σέγγεν ε, ρυθμίζονται σε διακυβερνητικό επίπεδο κατά το παρελθόν και τώρα έχουμε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ευρωπαϊκή διαχείριση του χώρου Σέγγεν. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίξει κεντρικό ρόλο, το είπε ο ίδιος ο Κάρλος, όσον αφορά την ετήσια και πολιτή αξιολόγηση και μέσω εκθέσεων που θα συντάσει. Νομίζω λοιπόν ότι η αλλαγή όσον αφορά τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση του χώρου Σέγγεν θα είναι κάτι θετικό. Θα ενισχύει τον χώρο αυτό της ελευθερίας που διαθέτουμε για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σχετικά με το μηχανισμό για την εισαγωγή ε, μεθοριακών ελέγχων είναι σημαντικό θέμα. Δεν θέλουμε να δούμε καταστάσεις όπως αυτές που είδαμε το 2011 όπου κράτη, μέλη, αυτοβούλος ε, επανέφεραν ελέγχους στα σύνορα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συμφωνία είναι καλή για τον χώρο Σέγγεν και ελπίζω ότι θα εθετηθεί η έκθεση άνευ προβλημάτων και από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών και από την Ολομέλεια στην επόμενη μήνυ Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Νταρόκα. Ευχαριστώ. Of course, first of all, I would like to appreciate immense work and patient. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κάλλος Κοέλιο, η τεράστια υπομονή του και τη Ρενάτε Βέμπερ που δεν είναι εδώ, θέλω να ευχαριστήσω. Πάνω από ένα χρόνο κουβεντιάζαμε τις προτάσεις. To introduce και προσπαθούμε να εισαγάγουμε μία ευρωπαϊκή αντί της προσεγγίσεως των κρατών μελών. Όμως και χτες είπα αυτά που θέλω να πω τώρα και στον τριμερή διάλογο. Θέλω να τα πω λεπτομερέστερα τώρα. Σε επίπεδο μελών της ΛΥΜΠΕ, της ομάδας μας, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε καμία από τις εκθέσεις. Θα αποφασίσουμε σε επίπεδο ομάδας την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι στεναρή θέση μας. Ήμασταν αρχικά για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Τροπολογία, αλλαγή του κώδικα των συνόρων και θέλαμε να υπάρξει και ένας μηχανισμός αξιολόγησης. Σχετικά με τις τροπολογίες, τις αλλαγές του κώδικα των, των συνόρων στην έκθεση Weber εκτιμούμε ότι υπάρχουν κάποια μέτρα διαφύλαξης διαδικαστικά. Όμως, όμως ακόμα πιστεύουμε ότι δεν μπορούν οι αλλαγές να είναι διακοσμητικής φύσεως. Διότι κατά στα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια, όπως είπε και ο Σέντσου, το απέδειξαν ότι χρειάζεται μια προσέγγιση ευρωπαϊκή. Και δυστυχώς απέτυχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επερασπιστεί την προσέγγιση της Ένωσης όπως έπρεπε. Όμως, παρόλα αυτά, κατά την άποψή μας, το Κοινοβούλιο έπρεπε να προχωρήσει στην εξέταση του θέματος. Uh, Γι' αυτό έχουμε αυτή τη θέση όσον αφορά τα προτινόμενα δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τη συμβιβαστική συμφωνία όσον αφορά την έκθεση Κοήλιο τώρα. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η αλλαγή της νομικής βάσης δεν ήταν η ενδεδειγμένη λύση και το άρθρο 77 θα ήταν η πιο ενδεδειγμένη νομική βάση. Δυστυχώ όμως η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου παρετήθηκε, τα παράτησε μάλλον, και έχουμε αυτή την κατάσταση. Η μεγαλύτερη μας ανησυχία είναι η μνήμα της παράνομης μετανάστευσης. Θα προστιμούσαμε να αναφέρονται μεταναστευτικές ροές η λέξη παράνομος, παράνομη να μην αναφέρεται. Αυτός είναι ο τελικός συμβιβασμός και είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το συμβιβασμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μοσχάμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια μικρή παρέμβαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Θέλω να πηχήσω αυτά που είπε η Επίτροπος Μάλστρομ εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξίσου ικανοποιημένη με σας. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα, να προχωρήσουμε πιο πέρα, να δείτε τι έγινε πριν από ένα χρόνο. Ήταν πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Είχαμε εντάσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και νομίζω ότι το τελευταίο χρόνο όλοι καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές και τώρα έχουμε δύο νομοθετικά κείμενα επί που πρέπει να μας ικανοποιούν. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, έχει βελτιωθεί ο μηχανισμός. Όπως είπε ο κ. Κοέλιο, έχουμε κατάλογο βελτιώσεων. Θα έχουμε ευρωπαϊκό μηχανισμό και για την αξιολόγηση Σέγγεν και για την επανεισαγωγή μεθοριακών ελέγχων εάν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στα σύνορα. Σίγουρα κάναμε ένα βήμα πρόοδου και πέρα από τις νομοθετικές προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει με την, α, ε, την ε, έκθεση. Η τρίτη έκθεση θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα και βάσει της εκθέσεως όλα τα θεσμικά όργανα θα έχουν πολιτική συζήτηση και θα υπάρχει και αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη. Thank uh, Εκθέσεις θα έρχονται μια φορά κάθε δύο χρόνια. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνω τη συζήτηση. Κύριε Κοέλιο, θέλετε να δευτερολογήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή και την υποστήριξή τους και θέλω να πω ότι καταλαβαίνω γιατί κυρία Ρανόκα δεν είναι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα. Θα προτιμούσαμε να έχουμε συναπόφαση. Και δεν μου αρέσει η διατύπωση που δεχτήκαμε χθε. Βέβαια, σε μια συμφωνία πάντα υπάρχουν κάποια σημεία που δεν μας αρέσουν πολύ. Για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, είχαμε ευθυγραμμιστεί με την ιδέα που είχαμε σχηματίσει στην Επιτροπή. Να μην επιτρέψουμε να βάλουμε τη λέξη παράνομη με άτομα. Σε κανένα σημείο του κειμένου δεν μιλάμε για παράνομους μετανάστες ή παράνομα άτομα. Η έκφραση όμως παράνομη μετανάστευση είναι στις συνθήκες και είναι πολύ δύσκολο για το Κοινοβούλιο να επιχειρηματολογήσει ε, ο, λέγοντας ότι είναι κάτι που πρέπει να διαγράψει. Το Συμβούλιο θα πει εντάξει, ας το διαγράψουμε πρώτα, ας διαγράψουμε αναφορά τη συνθήκη. Εν πάση περιπτώσει, πετύχαμε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Το Συμβούλιο δέχτηκε να μην βάλουμε μόνο την παράνομη μετανάστευση, όπως αναφέρει στις συνθήκες, αλλά να προσθέσουμε και όλα τα άλλα τμήματα της εντολής Frontex που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο να προσθεθούν. Είναι καλύτερο δηλαδή, καλύτερη κατάσταση. Κατανοώ τη θέση σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Ήταν πολύ καλή και συνεπής καθ' όλη τη διαδικασία, αλλά σας εκλυπαρώ να σκεφτείτε τι είναι καλύτερο να κολλήσουμε στο διακυβερνητικό μοντέλο αξιολόγησης που ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί ή να επιλέξουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση που εγκρίναμε και συμφωνήσαμε Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Ειλικρινά πιστεύω ότι αν τα συγκρίνουμε θα συμφωνούμε ότι όλα τα παρά τις, τα λάθη, τα προβλήματα το νέο σύστημα είναι πολύ καλύτερο από το παλιό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θα κυκλοφορήσει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, email, σύντομα προς τα μέλη, σήμερα ή αύριο. Θα συμπεριλαμβάνει το κείμενο των συμφωνιών και τη σύσταση του κυρίου Κοέλιο, προθεσμία για τροπολογίες θα καθοριστεί την επόμενη ως όριο, επόμενη τρίτη το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα το ταχύτερο δυνατόν μετά, ενδεχομένως 6 ή Ιουνίου στο Στρασβούργο νομίζω. Καλώς, άρα ολοκληρώσαμε τη συνεδρίασή μας, εκτός αν έχετε κάτι στα διάφορα, όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.